σαφή. Όταν ο κύριο εδώ που σα είπα με τον Μπέζ Πουλόβερ σα κουνεί στο χέρι, παρακαλώ να χαμογελάσετε. Περνάμε λοιπόν τώρα κυρίε και κύριοι στην ψηφοφορία. Και πριν περάσουμε στην ψηφοφορία έχω μία παράκληση ανακοίνωση. Παρακαλώ λοιπόν, Στο τελο των ε, ψηφοφοριών, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι ψηφοφοριε σα παρακαλώ για μικρό χρονικό διάστημα να παραμείνετε καθισμένοι γιατί έχω να σα κάνω μία σημαντική ανακοίνωση. Παρακαλώ λοιπόν στο τελο τη ε, ψηφοφορία μείνετε καθισμένοι πρέπει να σα κάνω μία σημαντική ανακοίνωση. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Ενιριάντα. Η συγγήτρια έχει το λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, λόγω ακριβώ τη οικονομική κρίση είχαμε το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι ένα ταμείο πάρα πάρα πολύ χρήσιμο, διότι έτσι μπορεί, μπορούν τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν αυτού οι οποίοι έχασαν τη δουλειά του κατά την κρίση. Ε, τώρα μπορούν αυτοί να καταρτιστούν, μπορούν ε, να έχουν καινούργιε δεξιότητε και έτσι να έχουν περισσότερε πιθανότητε πρόσβαση στην αγορά απασχόληση. Πρόκειται για ε, μια επένδυση όσον αφορά την απασχόληση, όσον αφορά το πώ οικονομικά βιώσιμα θα είναι αυτά όλα τα, άτομα. Οπότε παρακαλώ οι εθνικοί νομοθέτες να βοηθήσουν αυτού του είδους την κινητοποίηση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και κυρίως στα κράτη τα οποία έχουν τώρα τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι χρειάζεται κάποια αρρωγή, χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα της αγοράς απασχόλησης καλύτερη ε, προσβασιμότητα, χρειάζεται ένα διαφορετικό ήθος και θα πρέπει να υπάρξουν ενισχύσεις σε περιφερειακό επίπεδο επίσης. Οπότε, ό,τι συνάδει με τις διατάξεις που διέπουν το Ταμείο αυτό, θα πρέπει να καλυφθεί. Οπότε αυτό θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλη η εμπειρογνωμοσύνη. Παρακαλώ, υποστηρίξτε την εν τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Φαντάζομαι ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Τερμά συγχαρητήρια κυρία Νιδιάντα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Κίρτσου κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, ε, επίση ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Από ό,τι βλέπω ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία και η έκθεση αυτή εγκρίθηκε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα μικρό τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Οι φωτογράφοι δεν μπορούν να σας φωτογραφίζουν την ώρα που ψηφίζετε και είσαστε ασχολημένοι με την συσκευή ψηφοφορία. Κοιτάξτε, θα τελειώσουμε γρήγορα με τι ψηφοφορίε και σα κάνω την εξή πρόταση. Αν μετά παραμείνετε καθισμένοι, ε, θα μπορούν να κάνουν τι φωτογραφίε, ή μάλλον τώρα, τώρα να σα βγάλουν τι φωτογραφίε και μετά να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Συμφωνείτε τώρα να βγουν οι φωτογραφίε. Λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη να βγουν γρήγορα οι φωτογραφίες, παρακαλώ μείνετε καθισμένοι. Ε, και ρωτώ λέει ο πρόεδρος, εμένα θα με πάρετε φωτογραφία γιατί από ό,τι φαίνεται ο μόνος που δεν θα πάρετε φωτογραφία θα είμαι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, κυρίως γιατί αντέξατε και με πειθαρχία μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ε, ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μουρεσάν και εδώ ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γετενμέκη, ε, επίσης ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Περνάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Τάνκ. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Και περνάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Γκονζάλες Πόνς. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε και η τελευταία έκθεση. Σας παρακαλώ πολύ και πάλι για λίγο την προσοχή σας. Όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της 16 η Ιουλίου ο ε, συνάδελφος Ευρωβουλευτής Κόρβιν Μίκελ ε, προέβησε δηλώσεις ε, οι οποίες δεν συνάδουν με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ρατσιστική